του εσωτερικού κανονισμού 3 ε, και 4 του εσωτερικού κανονισμού έχει, έχει ε, επικυρωθεί ότι ε, ζήτησε επικύρωση της θητείας του ο Ευρωβουλευτής Κέντ Γιώχανσον από τις 21 Οκτωβρίου και ε, προτείνω να την δεχθούμε. Έχετε παρατηρήσει, αν όχι τότε επικυρώνεται η θητεία του κυρίου Γιώχανσον. Ο κύριος Ελί Χοουραού μου ανέφερε ότι παρετείται από Ευρωβουλευτής